Good afternoon, dear colleagues. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Δυστυχώς η Ολομέλεια δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Έχουμε την Ολομέλεια για ε, το από του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ από το σημείο που σταματήσαμε σήμερα το πρωί σημείο υπαριθμών 9. Θα θυμάστε ότι σήμερα το πρωί αναβάλαμε το σημείο 8, διότι η κυρία Γκάλ, η συγγήτρια για την ε, θεσμικέ πτυχέ τη προσχώρηση Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων, δεν είναι εδώ σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα περάσουμε στο σημείο 9. Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Schengen, SIS 1, συν, στο σύστημα πληροφοριών Schengen δεύτερης γενεάς, SIS-2. Τροποποίηση μιας προηγούμενης απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ε, του Συμβουλίου ε, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Κοέγιο. Το σημείο 10 αφορά στη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Schengen SIS-1 συν στο σύστημα πληροφοριών Schengen Δεύτερη γενεά και τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν και θα συζητήσουμε τα δύο αυτά θέματα από κοινού. Θα γίνει μια σύντομη συζήτηση για τις τροπολογίες που κατατέθησαν ε, στα δύο σχέδια εκθέσεων του κυρίου Κόεγη για το, η μετάβαση από το σύστημα πληροφωνών c ΣΥΣ1 στο σύστημα δεύτερης γενεάς, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 15 Μαρτίου έχουν κατατεθεί οκτώ τροπολογίες για κάθε μία από τις δύο εκθέσεις. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει γνωμοδοτήσει και για τις δύο ε, εκθέσεις αυτές και συντάκτης ε, και για τις δύο εκθέσεις αυτές είναι ο κύριος Άλβερο, ο οποίος είναι παρόν εδώ σήμερα συνεδρίαση. Ε, έχουν αποσταλεί οι τροπολογίες στα μέλη στις 26 Μαρτίου. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν τον κύριο Κοέγιο και στη συνέχεια, ως συνήθως, θα έχετε το λόγο και η Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να σας υπενθυμίσω ότι στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας θα ψηφίσουμε τα δύο θέματα αυτά, 27, Απριλίου και 27 και 28 Απριλίου. Σημειώστε λοιπόν ότι θα ψηφίσουμε 27 και 28 Απριλίου. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Κοέγιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς όλους όσους παρουσίασαν ανθρωπολογίες και πρωτίστως τον κύριο Άλβαρο. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τις γνωμοδοτήσεις του. Συμφωνώ με την γραμμή που ακολούθησε η Επιτροπή Προϋπολογισμών, ε, στην οποία αντικατοπτρίζεται και ο ο συμβιβασμός στο οποίο κατέληξαν το ΕΛΚ, οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι. Όλα αυτά φαίνονται και στις τροπολογίες στην Επιτροπή, που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού. Όσον αφορά τώρα στις τροπολογίες στην εκθεσή μου, έχω κάποιες ε, αμφιβολίες για τις τροπολογίες 17 και 18. Είμαι όμως διατεθειμένος να τις υπερψηφίσω. Τι συμβαίνει. Εγώ ανέκαθεν θεωρούσα ότι αυτή η νέα ομάδα διαχείρισης η οποία συστήθηκε για να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το, αυτό το Global Project Management Board θα πρέπει να είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα ασχολείται με θέματα τεχνικής φύσεως. Διαπίστωσα όμως ότι το Συμβούλιο έχει προβλέψει την διεύρυνση της συμμετοχής αυτής της συνεδριάσης σε πολλούς άλλους εμπειρογνώμονες, κυρίως από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν όντω ισχύει αυτό, συμφωνώ με ε, τη γραμμή του κυρίου Άλβαρο. Εάν θεωρούμε ότι θα έχουμε μια ομάδα περιορισμένη και τελικά είναι μια ομάδα η οποία ανοιχτεί για περιόριστο αριθμό μελών ε, ε, άλλων θεσμικών οργάνων, γιατί θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βρίσκεται στο περιθώριο. Έχουμε λοιπόν δύο επιλογές ή θα επανέλθουμε στο αρχικό σχέδιο, δηλαδή να έχουμε μια τεχνική ομάδα κλειστού χαρακτήρα ή αν ανοίξει θα πρέπει να ανοίξει για όλα τα θεσμικά όργανα και όχι μόνο για κάποια εξ αυτών. Αν και εγώ θα προτιμούσα το αρχικό μοντέλο μιας πιο τεχνικής ομάδας και πιο ειδικευμένης. Υπάρχουν επίσης οι προτάσεις ε, τροπολογίες ε, του συναδέλφου Ένσιο, του Σοσιαλιστικής Ομάδας. Εγώ έχω μόνο κάποιες ε, προτάσεις διορθωτικές. Ο συνάδελφος πρότεινε την διευκρίνηση των στοιχείων είναι μια απλή αλλαγή, η οποία είναι ευπρόσδεκτη, αλλά νομίζω πως το άρθρο 15 θα έπρεπε να είναι πιο καλό, πιο απλό, εάν ε, εκεί εισήγαμε και το 14. Αλλά είναι απλώς θέμα διατύπωσης. Απλώς ε, τη διαδικασία, διαδικασία της ψηφοφορίας θα ήθελα απλώς ε, να το προτείνω και ελπίζω πως και ο προτείνων τοπολογία θα συμφωνήσει. Πάντως θεωρώ ότι στη συμβαστική που επιτύχαμε με το Συμβούλιο σε σχέση με τις θεωρήσεις μακράς διαρκείας μια απόφαση που ήδη έχει αρχίσει να ισχύει στις 5 Απριλίου, υπάρχει μια δήλωση κοινή ε, και πρόθεση κοινή ότι δηλαδή προχωρούμε μέσα στο πλαίσιο του Σέγγεν ε, να έχουμε κοινά στοιχεία ε, στην περίπτωση που υπάρχουν περαιτέρω καθυστερήσεις στην έναρξη ισχύου του συστήματος. Τέλος, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν και σκεφτόμουν το συνάδελφο που έχει υποβάλει τροπολογίε, η μόνη που δεν μπορώ να δεκτώ είναι η 16, γιατί στο επίπεδο ε, που έχουμε στην αρχική πρόταση είναι πιο υψηλή η προστασία από αυτήν που θα είχαμε αν δεχτούμε την πρόταση 16. Δηλαδή, στην πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων, ε, με τις ε, συζητήσεις και με τις διαπραγματεύσεις που έχουμε, Θέλαμε να σβήνονται τα αρχεία στο τέλος ενός χρόνου. Κατά τη διάρκεια της συμβιβαστική ε, βρήκαμε μια προσωρινή λύση που έλεγε ένα χρόνο και το αργότερο τρία χρόνια μετά από τη δημιουργία του αρχείου. Άρα λοιπόν τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν αυτό το διάστημα. Η πρόταση τώρα του συναδέλφου Λουάν είναι να ξεπεραστούν και τα τρία χρόνια, πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πιο περίπλοκο από την ε, λύση που είχαμε αρχικά βρει και που κατά την άποψή μου είναι πιο αποδεκτή. Αυτή είναι λοιπόν η αντίδρασή μου σε σχέση με τις ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Thank you, Mr now before hearing την Προεδρία, την Επιτροπή, κυρία Άλβαρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω ότι η συνεργασία με τον κύριο Κοέλιο ήταν εξαιρετική. Συνεργαστήκαμε με εξαιρετικό τρόπο μέσω των Επιτροπών είμαστε μέλη αυτής εδώ της Επιτροπής και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί όσον αφορά τις τροπολογίες ακούσαμε την άποψή του. Θα ήθελα απλώς να επαναλάβω ότι οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί δεν έχουν σαν σκοπό να εμποδίσουν την ανάπτυξη του συστήματος SIS, αλλά να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα 80 εκατομμύρια που έχουν ήδη επενδυθεί στο πρόγραμμα αυτό και για το οποίο υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ερμηνείες θα οδηγήσουν σε επιτυχία. Γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν κάποιες, κάποια ερωτηματικά κάποιες στοιχές του προγράμματος. Συμφωνούμε λοιπόν και υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά τη γενική κατεύθυνση, αλλά θα ήθελα να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες. Ευχαριστώ. Η Προεδρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Κοέλιο και τον κύριο Άλβαρο οι οποίοι εξήγησαν πάρα πολύ καλά ε, τι περιλαμβάνουν οι τροπολογίες που κατέθεσαν. Από πλευράς ε, Προεδρίας του Συμβουλίου μπορούμε να πούμε εδώ στην Επιτροπή σας ότι η ευαισθησία των εισηγητών ε, στις ε, συναντήσεις που κάναμε στο παρελθόν ε, συνάδει με την ευαισθησία που έχει και η Προεδρία για τα θέματα αυτά στις διάφορες συζητήσεις. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι διαφυσβήτητα και το Συμβούλιο πάντα υποδέχεται ευπρόσδεκτα οτιδήποτε μπορεί να διασφαλίσει ότι θα έχουμε το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων όταν έχουμε ένα σύστημα πληροφοριών το Συμβούλιο σε ένα κείμενο το οποίο αφορά στη μετάβαση μεταξύ δύο στιμάτων ε, πληροφοριών και θα ε, θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε προστασία συνόρων και συνεργασία της αστυνομίας και των συνοριοφυλάκων σε καθημερινή βάση, ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει μία μετάβαση η οποία θα είναι εγγυημένη από όλες τις πλευρές. Επειδή ακριβώς λοιπόν υπάρχουν όλες αυτές οι εγγυήσεις στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάποια θέματα έχουν ήδη συζητηθεί στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να επιτύχουμε. Ε, πρόκειται για ένα σύστημα μετάβασης από το ένα σύστημα στο άλλο και το οποίο θα μας διασφαλίσει ότι θα μπορέσουμε να περάσουμε στο σύστημα δεύτερης γενεάς με όλες τις εγγυήσει για ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μια πτυχή που ανησυχεί ε, και προέκυψε από τις συζητήσεις που κάναμε στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Είναι το θέμα που αφορά στην τροπολογία 17, αυτό που σχολίασε και ο κ. Κοέλιο. Το η ομάδα διαχείρισης είναι μία ομάδα η οποία θα είναι ε, τεχνικού χαρακτήρα. Το μέγιστο όριο έχει κλείσει στο ε, κείμενο το οποίο συζητάμε στην ομάδα εργασίας, υπό την έννοια ότι μιλάμε για ένα κλειστό αριθμό 10 εμπειρογνωμόνων, από τους οποίους 2 μπορούν να προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 8 εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Και η μόνη εξαίρεση στον αριθμό της ομάδας εργασίας είναι η δυνατότητα, επειδή αυτοί οι εμπειρογνώμονες καθορίζονται από συγκεκριμένα κράτη-μέλη, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συνέχεια στην εργασία, να μπορεί να επιτρέπεται και η παρουσία της ε, Προεδρίας ε, ανα πάσα στιγμή, περιτροπής Προεδρίας. Ε, όπως σας είπα, ο μόνος στόχος είναι να διασφαλίσουμε τη συνέχεια των εργασιών. Από εκεί και πέρα, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να αμφισβητήσω την επιθυμία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρχει και συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Να σας πω όμως ότι εγώ ως υπεύθυνο στη μόνιμη αντιπροσωπεία για τα θέματα του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν, όχι από τεχνικής πλευράς φυσικά, δεν ε, πήγαινα συχνά σε αυτές τις συνεδριάσεις και εγώ δεν θα σας το συνιστούσα σε καμία περίπτωση γιατί είναι τόσο τεχνικού χαρακτήρα που δεν θα καταλάβετε και τίποτα. Από πλευράς ε, Συμβουλίου είμαστε βέβαιοι ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρίσταται ανα πάσα στιγμή και να ενημερώνεται όποτε υπάρχει ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτό έκανε και η Ισπανική Προεδρία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Είμαστε βέβαιοι ότι το έκαναν και οι Προεδρίες προηγούμενες περιπτώσεις και θα το κάνουν και οι μελλοντικέ Προεδρίες. Το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται. Αυτή η ομάδα όμως είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα εξαρτάται από μία από τις επιτροπές ε, που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα σχέδια για τα οποία είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολουθείται και η διαδικασία της επιτροπολογίας. Ε, αυτό που θα μπορούσα να σας πω λοιπόν με πάσα ειλικρίνεια είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει σεβασμό στην αναλογικότητα αν έχουμε παρουσία μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την ε, ομάδα. Να πω για άλλη μια φορά ότι χαίρομαι για τα όσα έχει κάνει ο κ. Κόαγιος στην εκθεσή του και Από πλευράς Προεδρίας, ε, με την επιφύλαξη βέβαια και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ε, να σας πω ότι έγιναν ε, πριν από λίγο διάστημα οι τελικές συνεδριάσεις για να δούμε τα αποτελέσματα της πρώτης δοκιμής και η Προεδρία και το Συμβούλιο μπορώ να σας πω ότι είναι αισιόδοξοι. Θεωρούμε ότι αυτό το milestone θεωρούμε ότι έχει ξεπεραστεί. Ε, Πρέπει να γίνουν κάποιες ακόμα τυπικές συνεδριάσεις, ε, κάποιες συνεδριάσεις σε ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και κάποιες επιτροπές υψηλού επίπεδου, αλλά είμαστε αρκετά αισιόδοξοι, θεωρούμε ότι αυτός ο κανονισμός ε, για τη μετανάστευση θα μπορέσει να υλοποιηθεί σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Προεδρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Καταρχήν ευχαριστώ την Επιτροπή Ελευθεριών για την ε, στάση της και στα δύο αυτά κείμενα. Θα κάνω πολύ σύντομα σχόλια. Πρώτον, όσον αφορά τη δυνατότητα που έχει το Κοινοβούλιο να βάλει στο αποθεματικό το προϋπολογισμό αυτό είναι κάτι που δεν θα το σχολιάσουμε. Θα ήθελα απλώς εκ μέρους Επιτροπής να πω ότι θα πρέπει η διαδικασία να είναι σαφής, να είναι αποτελεσματική, έτσι ώστε εάν υπάρξει ανάγκη να μπορέσουν να αποδεσμευθούν αυτά τα κονδύλια. Να μην υπάρξει δηλαδή διαδικαστικό πρόβλημα και εμπόδιο στην εξέλιξη του προγράμματος. Δεύτερον, όσον αφορά την ομάδα την GPND. Πρόκειται για μια τεχνική ομάδα, ομάδα εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει την Επιτροπή όσον αφορά την καθημερινή διαχείριση και επειδή μπόρεσα να συμμετάσχω σε κάποιες από τις συνεδριάσεις ομάδας αυτής, θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ τεχνικό ο τρόπος που εργάζονται. Αν δεν είναι κανεί εμπειρογνώμονα, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώ τι γίνεται στην ομάδα αυτή. Θεωρώ λοιπόν ότι αν ανοίξουμε τη συμμετοχή στι συνεδριάσει της ομάδας αυτής στα θεσμικά όργανα, θα χάσουμε, αν θέλετε, λίγο από την ε, αποτελεσματικότητα Πρόκειται για εμπειρογνώμονες, πρόκειται για ειδικού και δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι πρέπει να ανοίξουμε τη συμμετοχή. Όσον αφορά τις τροπολογίες 15 και 16, δηλαδή όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, η Επιτροπή θεωρεί ότι στη φάση που βρισκόμαστε δεν χρειάζονται επιπλέον άρθρα για την προστασία των δεδομένων, διότι μέχρι την μετανάστευση υπάρχει η Συμφωνία του Σέγγεν, που είναι, αν θέλετε, το πλαίσιο από εκεί και πέρα και όταν θα αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα η προστασία των δεδομένων και ο κανονισμός 45-2001 θα αρχίσει να ισχύει πλήρως και τα συστήματα, το κάθε ένα από τα συστήματα Μάλλον δεν θα συνεχίσω. Το Ζητώ συγγνώμη. Τροπολογία 16, λέει ο μιλητής, που αφορά Όπως και ο εισηγητής, η Επιτροπή θεωρεί ότι η διάταξη αυτή δίνει λιγότερη προστασία από αυτή που ήδη υπάρχει. Άρα δεν θα στηρίξουμε την τροπολογία αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Gracias a la Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι πλέον μπορεί να ξεκινήσει συζήτηση μεταξύ των μελών. Θέλει το λόγο και πάλι ο κύριος Άλβαρο καταρχάς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Συμβούλιο, την Επιτροπή για αυτά που είπαν όσον αφορά τις τροπολογίες. Πιστεύω ότι η 17 είναι μια τροπολογία στην οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε εάν η Επιτροπή και το Συμβούλιο συμφωνήσουν σε αυτό που είπε ο Κάρλος Κοέλιο. Είναι νομίζω πολύ λογικό να υπάρχει μία μικρή ομάδα εμπειρογνωμόνων και να συναντάτε για να εργάζεται και να μην γίνεται απλώς μία κοσμική συνάντηση. Πιστεύω πραγματικά ότι η τροπολογία αυτή θα μπορούσε να υποστηριχθεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, για την τροπολογία 18, το Συμβούλιο Διαχείρισης του Προγράμματος θα πρέπει να έχει έναν πολύ σαφή ρόλο. Παραδείγματο χάρη ενημερωτικό. Ε, εδώ περιμένουμε από την Επιτροπή ένα μήνυμα, αν ναι ή όχι, μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Τώρα, για την τροπολογία 15. Εγώ έχω διαφορετική άποψη από αυτό που μας παρουσίασε εδώ εκπρόσωπος της Επιτροπής. Αυτό που μας προτείνατε είναι ουσιαστικά ένα πακέτο μέτρων όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όπως ξέρετε υπάρχει και ένας άλλος κανονισμός του 2005 όσον αφορά τα προβλήματα σε θέματα ασφάλειας και θα πρέπει να δούμε αν στην αναθεώρηση αυτού του κανονισμού έχουν καλυφθεί τα σημεία αυτά που προτείνουμε με την τροπολογία 15. Αν όχι και αν δεν εφαρμόζεται εδώ ο κανονισμός αυτός, τότε η τροπολογία 15 θα πρέπει να παραμείνει. Εγώ περιμένω από την ε, Επιτροπή να μου πει αν και οι δύο κανονισμοί εφαρμόζονται και ισχύουν εδώ. Γιατί σε περίπτωση παραβιάσεων ε, και ελλειπούς προστασίας, εδώ πραγματικά δεν μπορούμε να καλυφθούμε μόνο από τον έναν κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Vreau să-mi exprim din nou satisfacția faptului că uh, lucrez cu domnul Este Σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη η συνεργασία με τον κύριο Κοέλιο και τον κύριο Άλβαρο. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά και το πρώτο που θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά όλα τα μέτρα που θέλουν να λάβουν. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν θα πετύχει ή θα αποτύχει αυτό το πείραμα. Μας λείπουν κάποια στοιχεία και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Συμφωνώ πολύ με τον κύριο Άλπαρο ότι δηλαδή η τροπολογία 15 που θα πρέπει να πάει στο άρθρο 14, όπως είπε και ο εισηγητής. Δεν πρέπει λοιπόν να βγει η τροπολογία αυτή, καθότι πρόκειται ένα επιπλέον μέτρο. Ένα επιπλέον μέτρο το οποίο έχει σαν σκοπό την καλύτερη προστασία των δεδομένων. Και αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το διέξοδο. No more colleagues. No more questions. Ζητάει κάποιο άλλος το λόγο. Όχι. Ωραία. Κύριε Κοέλιο, έχετε το λόγο. Ε... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα της τροπολογίας 17. Θα ήθελα να είμαι σαφής. Εγώ θα προτιμούσα την λύση μιας μικρής κλειστής τεχνικής ομάδας. Αυτή ήταν η ιδέα και έτσι ιδρύθηκε αυτή η ομάδα, GPMB. Θα ήταν πολύ καλύτερα αν από την αρχή η Επιτροπή είχε στηρίξει αυτήν την ομάδα, GPMB. Όμως, αυτό δημιουργήθηκε την τελευταία στιγμή και η ιδέα είναι να συμπεριληφθούν εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη και να σιγουρευτούμε ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο τεχνικό και πραγματογνωμοσύνης για το πρόγραμμα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν. Με την πρόταση που έχουμε εδώ και η οποία λέει ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει ο αριθμός των 10 στην ομάδα αυτή, GPMB, άλλα μέλη της Επιτροπής μπορούν να συμμετάσχουν με δικά τους έξοδα. Καταλαβαίνω τι λέει το Συμβούλιο. Θέλει να διευρύνει σε μέλη της Επιτροπής αλλά και σε εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Στο κείμενο εργασίας του Συμβουλίου διευρύνεται λοιπόν η συμμετοχή στην ομάδα αυτή. Και δεν θεωρώ ότι αυτή η πρόταση είναι πολύ καλή. Εγώ προτιμώ την λύση του κυρίου Άλβαρο γιατί να υπάρχουν μέλη της Επιτροπής, μέλη και εμπειρογνώμονες από τα κράτη και όχι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Δεν καταλαβαίνω. Κατά την άποψή μου λοιπόν υπάρχουν δύο λύσεις που μπορούμε να δεχτούμε. Είτε θέλουμε να μειωθεί αυτή η ομάδα σε δέκα μέλη τεχνικούς δηλαδή, εμπειρογνώμονες και κανέναν άλλο, είτε εάν διευρύνουμε τη συμμετοχή και συμπεριληφθούν και μέλη της Επιτροπής, Υπάρχουν επίσης εμπειρογνώμονες από το Συμβούλιο και από τα κράτη-μέλη, γιατί όχι και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε λύση. Μπορώ να προετοιμάσω μια συμβιβαστική λύση, αν θέλετε, όπως ε, άκουσα να προτείνει ο συνάδελφος, μπορώ να προετοιμάσω μια άλλη πρόταση, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει εκτός αυτής της ε, ομάδας. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο σχόλιο από πλευράς Προεδρίας ή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλετε να προσθέσετε κάτι μετά από τα συμπεράσματα του εισηγητή, του κ. Κόλλιο. Όχι. Ωραία. Να υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ 27 και 28 Απριλίου. Κύριο Άλβαρο, ευχαριστώ. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ μία απάντηση στην ερώτηση που έθεσα για την τροπολογία του κυρίου Εντσίου. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι ίσως απορρίψει αυτή την ε, τροπολογία και χρησιμοποιήσει ως αιτιολόγηση την ε, ε, οδηγία 9546. Αν όμως γνωρίζω καλά τα πράγματα, δεν υπάρχει κάτι στο 9546 που να αναφέρεται στην ε, ε, παραβίαση αυτών των όρων, όπως ε, είναι και η τροπολογία του κ. Έντσιου. Ίσως δεν γνωρίζω καλά τα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν κάποιες απαντήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο υπόσχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα απαντήσει στην ερώτηση του κ. Άλβαρο. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω την απορία του κυρίου Άλβαρο. Παρ' όλα αυτά θα το έθετα διαφορετικά εγώ. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόκειται σε υποχρέωση επίπεδου ασφάλειας εξαιρετικά υψηλού. Δηλαδή, ένα επίπεδο το οποίο απορρέει όχι από τον κανονισμό, αλλά από μία απόφαση συλλογική της Επιτροπής. Είναι υποχρεωμένη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει στους φορείς, τους οποίους αναθέτει αυτά τα, αυτές τις αποστολές, ένα πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας. ένα επίπεδο που πραγματικά φτάνει στο ύψιστο, στο βέλτιστο αν θέλετε επίπεδο ασφαλείας. Με αυτό λοιπόν ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό και μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, το υπαριθμό 11 στην ημερήσια διάταξη. Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Και πάλι συγκητής ο κύριος Κοέλιο. Θα ακούσουμε όμως μια σύντομη παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την τροπολογία που προτείνεται για, την για τον οργανισμό ε, βάση και τις επικαιροποίησεις που πρέπει να γίνει για τη συνθήκη της Λισαβόνας και τις επικαιροποίησεις που έχει ζητήσει το Συμβούλιο. Θα ακούσουμε λοιπόν τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά το Συμβούλιο και στη συνέχεια θα μιλήσει και ο εισηγητής, ο κύριος Κοέλιο και οι λοιποί συνάδελφοι που θα θέλουν το λόγο. Η Κομισιόν παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais, je vais très rapidement présenter. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας παρουσιάσω σύντομα την τροποποίηση του κανονισμού για τη δημιουργία ενός οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφορικών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Ο πυρήνας της αποστολής αυτής, αυτού του οργανισμού που προτείνεται είναι να κάνει ε, δραστηριότητες λειτουργικές διαχείρισης για διάφορα συστήματα πληροφορικής όπως το SIS-2 για το οποίο μιλήσαμε, το FIS και το EuroDAC. Και στο μέλλον και με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν τα κατάλληλα νομικά μέσα θα μπορούσε επίσης ο οργανισμός να ασχοληθεί με την ανάπτυξη άλλων συστημάτων πληροφορικής στον τομέα της δικαιοσύνης της ασφάλειας και της ε, ελευθερίας. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο για την πρόταση που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2009 γίνανε στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση και ε, στο πλαίσιο των προτάσεων που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο, θα πρέπει να σα πω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Υπουργών τι υποστηρίζει τι προτάσει αυτές. Και αυτό γιατί α, με την έναρξη ισχύω τη Λισαβόνα. οι δομή σε πυλώνε που υπήρχε προηγούμενα ε, καταργήθηκε. Ε, και ως εκ τούτου η πρόταση για μια πράξη του τρίτου πυλώνα, γιατί πρόκειται για ένα πακέτο που αποτελείται από μια πράξη για τον πρώτο πυλώνα και μια πράξη για τον τρίτο πυλώνα, αυτή η πρόταση λοιπόν του τρίτου πυλώνα θεωρήθηκε πλέον ε, πεπερασμένη. Ενώ η πρόταση κανονισμού που αφορούσε τις δραστηριότητες του πρώτου πυλώνα έμεινε επιτάπητος. Οπότε η Κομισιόν χρειάστηκε να αποσύρει τον τρίτο πυλώνα στην ανακοίνωση Omnibus που αφορούσε την έναρξη ισχύω τη συνθήκη Λισαβόνα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με τη νέα συνθήκη η Ένωση έχει μια νέα αρμοδιότητα για να φτιάξει αυτή την επιρρήση των οργανισμό αλλά και όλε τι διατάξει που αφορούν τη λειτουργία του και αυτά όλα σε μια μόνη πράξη. Και αυτό και έκανε η Κομισιόν παρουσιάζοντα στι 19 Μαρτίου μια νέα πρόταση που στην ουσία είχε ω αποτέλεσμα να ενσωματώσει στην πρόταση κανονισμού στην πρώην δηλαδή, στον πρώην δηλαδή πρώτο πυλώνα τις προτάσεις που ήταν ήδη πεπερασμένες από το τρίτο. Να κάνει δηλαδή και μια καλλιντική, ε, όπως από την αποκαλώ εγώ, περιποίηση των πράξεων με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Να προσαρμόσει δηλαδή τις νομικές βάσεις. Ήταν τεχνικές παρεμβάσεις δηλαδή αποκλειστικά. Αυτά εστάλησαν και στα Εθνικά Κοινοβούλια και είμαστε σήμερα εδώ, ελπίζω, σε ένα πνεύμα εξαιρετικής συνεργασίας για να τα συζητήσουμε. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου θα είναι φυσικά κρίσιμος για τη δημιουργία αυτής της, του, του οργανισμού, αλλά και στην λειτουργία του, γιατί το Κοινοβούλιο θα είναι και η Δημοσιονομική Αρχή και η Ελεγκτική Αρχή για αυτό το νέο οργανισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Η Προεδρία θέλει να παρέμβει, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ να προσθέσω και πολλά σε αυτά που μόλις ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, θα ήθελα να πω λίγο εδώ στην Επιτροπή πώς έχει η κατάσταση και τι έχουμε επιτύχει σε προσωρινό χαρακτήρα ε, πάντα, γιατί μόλις πέντε συνεδριάσεις έχουν γίνει στην αρμόδια ομάδα εργασίας της ε, ε, του Συμβουλίου. Συγγνώμη. Υπάρχουν τρία ουσιαστικά θέματα, τα οποία λόγω της δυσκολίας του θέματος δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμα. Ε, το μοντέλο που θα πρέπει να έχει αυτός ο οργανισμός ε, προτείνονται δύο εναλλακτικές λύσεις. Η μία είναι μια κεντρική πρόταση όπως ήταν στο αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, υπάρχει και μια συγκεκριμένη λογική φυσικά και τη διέπει και υπάρχει και μια αποκεντρωμένη πρόταση με διάφορες τεχνικές πτυχές. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν ε, κάποιες τεχνικές έδρες αποκεντρωμένες και μια γενική έδρα. Ε, το σκεπτικό είναι να επιτρέπεται αποκέντρηση για λόγους ασφαλείας. Όλοι οι τεχνικοί φυσικά μπορούν να προασπίσουν αυτή τη δυνατότητα. Η αποκέντρωση δηλαδή μόνο των εδρών όπου υπάρχουν ε, αντίγραφα ασφαλείας, backup. Από πλευράς Προεδρίας δεν μπορούμε να πούμε ότι τίνουμε προς τη μία ή την άλλη λύση, γιατί η συζήτηση στο Συμβούλιο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει και ένα ακόμα σημείο αρκετά διαφιλονικούμενο, το οποίο προέκυψε κατά τις συζητήσεις. Επειδή πρόκειται για μία πρόταση που έχει την διάσημη ε, μεταβλητή γεωμετρία και έχουμε συμμετοχή κάποιων κρατών μελών στα συστήματα πληροφοριών που θα αφορούν στον οργανισμό, είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα δικαιώματα ψήφου, για το διευθυντή του οργανισμού ε, και την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ε, ξέρετε ότι αυτά είναι πολύπλοκα διότι Ερίζουν οι απόψεις στο θέμα αυτό ε, ως προς το ΣΥΣ, ε, το ΒΙΣ, το Eurodac ε, για, από πλευρά κρατών μελών. Υπάρχει κατά τρίτον και ένα ακόμα θέμα το οποίο δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα από την πλειονότητα των κρατών μελών και αυτό είναι η τροποποίηση που αποφασίστηκε βάσει της αρχικής πρότασης που αφορά την ίδια τη δομή του οργανισμού, όχι το μοντέλο των εδρών που συζητήσαμε πριν, αλλά την ίδια του τη δομή τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι ίσως θα πρέπει να ενισχυθεί η δομή του οργανισμού πέραν του Διευθυντή και του Διοικητικού Συμβουλίου με έναν ε, ε, αξιωματικό υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων, έναν αξιωματικό υπεύθυνο ασφαλείας για τα συστήματα πληροφοριών και κάποιον ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τα ε, δημοσιονομικά και λογιστικά θέματα. Αυτά αρχικώς είχαν θεωρηθεί καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και η πρόταση κάποιων κρατών μελών, ε, η οποία υποστηρίζεται από αρκετού στην ομάδα εργασία, είναι αυτές οι τρεις κατηγορίες να αποτελούν τμήμα της ε, ίδιας της δομής, ε, λόγω της σημασίας των τριών θεμάτων που μόλις σας ανέφερα. Αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους για συζήτηση. Πρώτον θα ακούσουμε τον εισηγητή, τον κύριο Κοέλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θυμίσω πως αυτή είναι μια υπόθεση την οποία θα πρέπει να ρυθμίσουμε με συναπόφαση. Είναι μια από τις σημαντικότερες ε, αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου που ο ρόλο μας είναι ευξημένος και θα πρέπει να λειτουργήσει όχι μόνο στην έγκριση του νομικού πλαισίου αλλά και στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων αυτού του οργανισμού. Θα ήθελα επίσης να θυμίσω ότι ακόμα δεν ξεκινήσαμε την εργασία μας με τους shadows για τις προτάσεις γιατί περιμέναμε αυτή την πρόταση της Κομισιόν γιατί με την έναρξη της ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας έπρεπε να γίνουν ε, αλλαγές όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που μας είχε προηγουμένως παρουσιάσει. Και η Κομισιόν ε, κατέληξε μετά από διάφορες συζητήσεις ε, και επέλεξε μάλλον την πρόταση, την, μάλλον την πρόταση υποβολής ενός ενιαίου κειμένου, μιας πρότασης κανονισμού σε σχέση με τις απορίες που υπάρχουν, τις αμφιβολίες που υπάρχουν, αυτές υπάρχουν γιατί δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη σε όλα τα συστήματα και ορισμένα κράτη-μέλη ε, συμμετέχουν μερικώς. Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα νομικής ε, ασφάλειας που τίθεται εδώ. Και γι' αυτό το λόγο κύριε Πρόεδρε θα σας στείλω μια επιστολή από μέχρι αύριο, ώστε θα ζητήσω με αυτήν η Επιτροπή μας να συμβουλευτεί την νομική υπηρεσία για να μας δώσει μια γνώμη για το ποιο είναι το καλύτερο, ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Να έχουμε δηλαδή ένα μόνο νομικό μέσο για τη ρύθμιση όλων αυτών των διαφορετικών θεμάτων όπου η συμμετοχή των κρατών μελών είναι διαφορετική. Έχουμε λοιπόν το Βρεντάκ, το ΒΙΣ και το ΣΥΣ και όπως ήδη υπόθηκε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν και άλλα, πρόκειται μάλλον για τη διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων. Και ξέρετε ότι για το Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό η απόδοση, η ανάθεση μάλλον νέων αρμοδιοτήτων σε αυτό τον οργανισμό να γίνεται μέσω νομοθετικής, της νομοθετικής οδού. Δηλαδή να μην είναι δυνατόν με κανένα τρόπο τα όργανα του οργανισμού να διευρύνουν τις αρμοδιότητες αυτού του οργανισμού στις πλάτες του αρμόδιου οργάνου, δηλαδή στις πλάτες του Κοινοβουλίου χωρίς την έγκριση δηλαδή του Κοινοβουλίου. Η Προεδρία μόλις μας θύμισε δε κάποιες λεπτομέρειες και εγώ θα ήθελα να πω πως ε, υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία είναι ευαίσθητα. Το πρώτο είναι το προφίλ, δηλαδή να ξέρουμε αν εμείς θα θέλουμε να έχουμε κεντρική διαχείριση όπως έχουμε αυτή τη στιγμή στο ΣΥΣ1 ή αν όπως κάποιοι υποστηρίζουν να έχουμε μια αποκεντρωμένη διαχείριση στα διάφορα κράτη-μέλη. Το θέμα της τοποθεσίας. Επίσης υπάρχουν διάφορες υποψηφιότητες, Γαλλία και Εστονία. Είναι βέβαιο πως πρόκειται για ένα θέμα που εν γέννη αποφασίζεται σε επίπεδο του Συμβουλίου, επειδή είμαστε στην απόφαση, αν αυτή η απόφαση, απόφαση ε, οδηγήσει σε διαφορετική σε διαφοροποίηση του προφίλ λειτουργία του οργανισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να μείνει εκτό αυτή τη συζήτηση. Το θέμα επίση είναι τη συμμετοχή των κρατών μελών σε σχέση με μάλλον ανάλογα με την συμμετοχή του σε κάθε ένα από τα συστήματα, όπω είπα και πριν. Έπειτα, αποσαφήνιση των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων αυτού του οργανισμού το θέμα της ε, ε, ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των στοιχείων, προστασία των στοιχείων δηλαδή, των δεδομένων. Και ε, στη συνέχεια η ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων που είναι κάτι το οποίο ζητάμε διαρκώς εδώ και χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Ισπανικής Προεδρίας θα πρέπει να αναφερθούμε σε πρωτοβουλίες που ήδη έχουν ξεκινήσει σε επίπεδο Συμβουλίου για να δημιουργηθεί ένας ε, υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή υπεύθυνο ασφάλειας δεδομένων στο κατάλληλο επίπεδο και να έχει στη διάθεσή του και τα απαραίτητα μέσα να, ενισχύσει το επί... να αυξήσει το επίπεδο μάλλον προστασίας των δεδομένων. Το Κοινοβούλιο σε όλα αυτά θα πρέπει να συμμετέχει συνοδεύοντας και ελέγχοντα τα όργανα, τα διοικητικά αυτού του οργανισμού. Αυτά είναι λοιπόν τα επτά πιο σημαντικά θέματα, πιο λεπτά ζητήματα από τον οποία θα χρειαστεί να λάβουμε θέση και το έγγραφο που μας παρουσιάζει η Κομισιόν το είδαμε τώρα και τώρα θα συνεργαστούμε με τους σκιώδεις συζητητές ώστε η Επιτροπή μας να μπορέσει σύντομα να ενημερωθεί για αυτό το ευρύ σύνολο προτάσεων και να μπορέσει να συναποφασίσει με το Συμβούλιο. Γιατί, επαναλαμβάνω, έχουμε ε, σημαντικό ρόλο καθώς πρόκειται για συναπόφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κόλλιο. Η κυρία Λάτφορ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για όλες τις παρουσιάσεις και αυτή που μας έκανε ο εισηγητής μας, του οποίου οι παρατηρήσεις καλύπτουν ένα τμήμα αυτών που ήθελα να ρωτήσω και αφορούσαν την παράταση της εντολής του οργανισμού για να καλύψει και άλλα συστήματα και άλλες βάσεις δεδομένων. Ο εισηγητής επεσήμανε ότι δεν μπορεί να επεκταθεί θα ήταν απαράδεκτο να επεκταθούν οι αρμοδιότητες χωρίς να περάσουν από το συνομοθέτη, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης την εξή ερώτηση. Έχουμε καμία εικόνα, κανένα εναλλακτικό σενάριο για τις άλλες βάσεις δεδομένων που θα προσθεθούν. Ξέρω ότι η Επίτροπος Μάλστρομ, η οποία είναι υπεύθυνη για το θέμα, μίλησε σε μένα και ίσως και σε κάποιους άλλους στη διάρκεια της ακρόασης και αναφέρθηκε σε μία ε, αναθεώρηση της κατάστασης για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού οδεύουμε για τη συλλογή δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' εμέ αυτό θα πρέπει να καλύπτει και τις εσωτερικές βάσεις δεδομένων. Ε, τα τελευταία πέντε χρόνια υπήρχαν αρκετές δυνατότητες, παρουσιάστηκαν αρκετές ιδέες, ε, θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια που συζητούσαμε μία αποκεντρωμένη βάση δακτυλικών αποτυπωμάτων που στη συνέχεια βέβαια έγινε μία ιστορία τρόμου. Ε, υπήρχε και απόφαση Ντεπρούν για την ανταλλαγή δεδομένων, ε, κατά πόσον αν αρχίσουν να ανταλλάσσονται τα δεδομένα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κατά πόσον υπόσχεση της Επιτρόπου Μάλστρομ να δούμε λίγο πώς έχει η κατάσταση και έναν οδικό χάρτη αναπτύσσεται αυτός ο οδικός χάρτης. Ποια είναι τα όρια της συλλογή δεδομένων σε, ε, ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να το ξέρω φυσικά, πιστέψτε με, και στη χώρα μου αυτό. Και πότε θα αρχίσουν τα πράγματα να σταματήσουν να είναι απλώς οικοασίες και να υλοποιηθούν, να είναι συγκεκριμένα σχέδια. Και αυτά τα συγκεκριμένα σχέδια θα τα μάθει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί στο παρελθόν διαπιστώσαμε, ε, για παράδειγμα με τα πιλωτικά προγράμματα που ανέφερε ο κύριος Κοέλιο, ότι είναι απλώς υποσημειώσει στον προπολογισμό και εμεί ε, διαπιστώνουμε μόνο στο σχέδιο προπολογισμού στις υποσημειώσεις τι σχέδια υπάρχουν για νέες βάσεις δεδομένων. Σε ποιο σημείο λοιπόν θα ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο συγκεκριμένη για τα μελλοντικά τη σχέδια, ώστε να μην βλέπουμε μόνο τα θέματα της προστασίας δεδομένων, αλλά και τι δυνατότητα σε επέκταση της εντολής αυτού του οργανισμού μπορούμε να έχουμε. Ευχαριστώ κύριε Λάτφορτ. Ο κύριος Άλμπερτ. Ευχαριστώ. Κατά την άποψή μου, Υπάρχουν τρία ενδιαφέροντα σημεία και σημαντικά για μένα. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρει το θέμα της προστασίας των δεδομένων που θα πρέπει να μπει στις αρμοδιότητες αυτού του οργανισμού δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει απλώς ένας εσωτερικός, ε, αν θέλετε, έλεγχος της προστασίας των δεδομένων. Αυτό δεν αρκεί κατά την άποψή μου και αυτό το υπογραμμίζω. Δεύτερον, το κόστος. Αναρωτιέμαι, αυτά τα 170 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται εδώ, αν δικαιολογούνται. Μιλάμε για μια υπηρεσία πληροφορικής, υπάρχει όλο το τεχνικό κομμάτι, αλλά θεωρώ ότι είναι υπερβολικό το ποσό. Δηλαδή η ανάπτυξη αυτών των διαδικασιών θα πρέπει σαφώς να λάβει υπόψη και τη δυνατότητα να αποφύγουμε επικαλύψεις, να μην υπάρξουν προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει κάπου αλλού Δηλαδή, σκοπός μας είναι αυτή η τεχνική, αν θέλετε, δουλειά να γίνει όταν και εφόσον και μόνο επειδή είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει κάπου αλλού. Αναρωτιέμαι λοιπόν αυτό το ποσό των 170 εκατομμυρίων ευρώ δικαιολογείται εδώ. Τρίτο σχόλιο. Οι αρχές προστασίας των δεδομένων και οι κανονισμοί που υπάρχουν. Βλέπω το σημείο 11, στην ευτολογική σκέψη 11, κάτι το οποίο δεν μου φαίνεται καθόλου δεσμευτικό. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα αυτό της προστασίας. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεκτημένο όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και αυτό που λέμε εμείς εδώ είναι μια ουσιαστικά τεχνική επεξεργασία των δεδομένων τίποτα δεν μου φαίνεται δεσμευτικό και θα πρέπει σαφώς να αποφύγουμε αυτή η τεχνική, αν θέλετε, συγχώνευση, ε, επεξεργασία, να μην λάβει υπόψη τις ε, δυνατότητες συνέργειας ε, και να δημιουργήσουμε προβλήματα μη συμβατότητας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την διαλειτουργικότητα και το διεπιχειρησιακό χαρακτήρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω, Δεν βλέπω κανέναν άλλο να ζητά το λόγο. Ωραία, λοιπόν. Η Κομισιόν θέλει κάτι να απαντήσει στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις που αφορούσαν το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο άρθρο 25 που είναι και λέει σαφώ ότι ο κανονισμός 47 του 2001 είναι ο ισχύων με όσο αυτό σημαίνει συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητα του DPS, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτή Προστασίας Δεδομένων. Δεν πιστεύουμε στο κείμενο αυτό πως ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθούν ειδικά άρθρα τα οποία θα παρέθεταν ή θα αντέγραφαν τι γενικέ διατάξει που ισχύουν στον κανονισμό 45 2001. Γι' αυτό θα πρέπει να, να έχουμε υπόψη μας ότι όλα αυτά ήταν ε, μια τεχνική αλλαγή, μια ε, πρόκειται για κάτι που πρέπει να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, μέσα στο πλαίσιο νομικών μέσων που υπάρχουν. Ο προπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ είναι ένας προϋπολογισμός τριετής και συμπεριλαμβάνει και εν μέρη τις εγκαταστάσεις. Αντίθετα, αυτός ο οργανισμός δεν έχει άλλη δραστηριότητα από αυτήν που συγκεκριμένα προβλέπεται από αυτό το νομικό μέσο ή που θα του ανατεθεί από επιπρόσθετα νομικά μέσα. Και εδώ μπορώ να επαναλάβω τα όσα είπα στις αρχικές μου παρατηρήσεις, ότι δηλαδή κάτι τέτοιο θα σήμαινε ένα συγκεκριμένο νομικό μέσο που θα δίνει στον οργανισμό τέτοια νέα συστήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος παράκαμψης, θα έλεγα, του νομοθέτη. Νομίζω ότι απάντησα στα υπόλοιπα. Ξέχασα ίσως την κυρία Λάτφορντ. Αυτό δηλαδή για το οποίο δεσμεύθηκε η Επίτροπος Μάλστρομ. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία και η κυρία Μάλστρομ θα ανταποκριθεί στις ε, υποσχέσεις της, στις υποχρεώσεις της όταν προχωρήσει η διαδικασία. Όσον αφορά στα επιπλέον συστήματα, χρειάζεται εδώ μια ξεχωριστή νομική βάση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Προεδρία θέλει να πει κάτι ακόμα. Άντε τότε πάλι εσείς κύριε Κοέλιο, ως εισηγητής για να κλείσετε τη συζήτηση. Ο τίποτα ιδιαίτερο δεν έχω να πω πρόεδρε, να θυμίσω μόνο στη Βαρόνη Λούτφορτ ότι μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπω ο οργανισμός, η εντολή μάλλον αυτού του οργανισμού δεν θα, είναι, δεν θα λέει ότι είναι ο τελικός καταναλωτής των πληροφοριών. Δηλαδή, ο ίδιος ο οργανισμός δεν θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία, στα δεδομένα. Θα παρέχει τα εργαλεία ώστε να μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Και έτσι ώστε να αραίουν φυσιολογικά, όπως είπε η Κομισιόν σωστά, 24 ώρες, 24 ώρο και 365 μέρες το χρόνο. να ρέουν οι πληροφορίες, δηλαδή ώστε κάθε αστυνομικός να είναι σε θέση να ελέγξει το σύστημα, να το ρωτήσει και να έρχει σύντομα τις απαντήσεις. Ε, μιλάμε για δευτερόλεπτα. Πρέπει λοιπόν να αναζητεί τις τεχνικές λύσεις ώστε να μπορεί να παρέχει μια καλή υπηρεσία, γρήγορα, με ένα ψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. <laughs> Αλλά ε, δεν είναι ζωτική σημασία να γνωρίζει το περιεχόμενο των πληροφοριών αυτών. Οπότε ορισμένοι από τους φόβους της Βαρόνες Λάτφορντ αν τα πράγματα λειτουργήσουν σωστά, όλα αυτά δεν είναι δικαιολογημένα, δεν στέκουν αυτοί οι φόβοι. Φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει μέσω νομικών μέσων ότι θα λειτουργούν όλα αυτά ομαλά. Μιλάμε για Ευρωπαϊκό Οργανισμό και ο κανόνας του Ευρωπαίου Επόπτη για τα στοιχεία ισχύει και δεν έχω άλλα τίποτα να πω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Λούτφορντ, συγγνώμη Πρόεδρε, επανέρχομαι γιατί και ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτή την παρατήρηση. και φυσικά το γνωρίζω ότι θα διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων, δηλαδή θα παρέχει μια κοινή πλατφόρμα, μια κοινή βάση. Και Βεβαίως, όταν αρχικά έγινε η πρόταση αυτή, τεχνική διαλειτουργικότητα σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάρχει ανταλλαγή ανάμεσα στις διάφορες βάσεις δεδομένων. Από την άλλη όμως πλευρά νομίζω ότι η ίδια ύπαρξη μια κοινή κεντρική ενό κοινού κεντρικού οργανισμού διαχείρισης και μια κοινή τεχνική πλατφόρμα, ενώ δεν σημαίνει αυτομάτως βέβαια ότι θα υπάρχει διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων και κοινή πρόσβαση στις πληροφορίες κτλ. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε το νου μας να μην λειτουργήσει ως μια βάση για μια προϋπόθεση ότι τώρα που υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία είναι ευκολύτερο να προστίθενται νέες ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων γιατί αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια οκνηρία και να, γι' αυτό να έχουμε το νου μας να μην ε, φτάσουμε σε τέτοιο σκεπτικό. Ότι είναι δηλαδή ένα μικρό βήμα για τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων. Σας ευχαριστώ κυρία Λούτφορτ. Κύριε Κουαλιό, έχετε να πείτε και τίποτα. Εγώ νομίζω πως η Βαρόνη Λούτφορτ και εγώ είμαστε στην ίδια γραμμή, στο ίδιο μήκο κύματος νέα λειτουργικότητα για αυτή τη νέα υπηρεσία θα πρέπει να δίνεται μέσω μιας νομικής πράξης, δηλαδή μια μέσω συναπόφαση με το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς στη διατύπωση αυτού του κειμένου ότι δεν πρόκειται να υπάρχουν νέες λειτουργίες, ούτε νέες βάσεις δεδομένων, ούτε νέες αρμοδιότητες, εκτός του νομικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει νομικό πλαίσιο που εγκρίνεται με τη συναπόφαση και με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Είναι κάτι το οποίο τόνισα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο και οι δύο θεσμοί γνωρίζουν ε, τι πιστεύει το Κοινοβούλιο περί όλων αυτών και πιστεύω ότι είναι ε, σύμφωνοι μαζί μας και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εγκρίνουμε στην εντολή αυτής της αυτού του νέου οργανισμού κάτι τελείως ξεκάθαρο ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε πειρασμοί ή κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε κύριε Κουέλιο. Κλείνουμε λοιπόν τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν στο σημείο 12 το οποίο θα εξετάσουμε από κοινού με το 13. Γιατί και τα δύο σχετίζονται με το PNR τους φακέλους PNR. Έχουμε την κυρία Ιντβελτ, που είναι η συγκίτρια για τις δυο αυτές εκθέσεις. Το 12 αφορά την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών από τους αερομεταφορείς στην στελωνικές υπηρεσίες της Αυστράλης και η 13 αφορά την συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ για την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών από τους αερομετωφερείς στο Υπουργείο Ιστορικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος εδώ είναι να έχουμε σήμερα μια ανταλλαγή απόψεων ώστε θα ζητήσω πρώτα στην εισηγήτρια κυρία Ιντφελτ να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. και τα μηνύματα που σκοπεύουν να υποβάλουν οι πολιτικές ομάδες στην επόμενη Λομέλεια την, ε, τον Απρίλιο. Έπειτα θα ακούσουμε την, την Κομισιόν, την Προεδρία και <coughs> αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας έρθουν θα δώσουμε το λόγο και στους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών των Ευρωπαίων Εκπροσώπων Προστασίας Στοιχείων. Α, όχι δεν θα έρθουν από ό,τι μου λένε. Είχαμε προβλέψει τον κύριο Χάσκινς και τον κύριο Μπουλγαρέλη που, θα... που θα ε, αντιπροσώπευαν την ε, Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων αλλά δεν θα έρθουν. Κύριε κυρία Ιντεφέλτ. Σύντομα κύριε Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε το θέμα αυτό. Θα σας δώσω λοιπόν μια σύντομη παρουσίαση για να σας υπενθυμίσω εάν δεν θυμάστε και να στηρίξουμε τις δύο μεγάλες συμφωνίες με την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων Σαν εισηγήτρια είχα προτείνει να αναβάλουμε καταρχήν την ψηφοφορία, καθότι πάντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τοποθετηθεί αρνητικά. Και έτσι να αποφύγουμε την απόρριψη αυτών των ε, συμφωνιών, κάτι που θα δημιουργήσει σύγχυση και για τους ε, επιβάτες και για τις ε, αεροπορικές εταιρείες. Να προετοιμάσουμε λοιπόν προτάσεις για μία προσέγγιση με συνοχή, μία κοινή ε, στάση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα αυτό όσον αφορά τη συμφωνία με τον Καναδά που έχει ε, λήξει και την ε, πιθανή αντιμετώπιση του θέματος αυτού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία σειρά μέτρων η οποία να μπορεί να ισχύσει και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των ε, συμφωνιών με άλλες χώρες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν για την πολύ φιλική και ανοιχτή του στάση. Επίσης το ίδιο θα έλεγα και για την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Εδώ υπάρχει σαφώς ε, μια συνεργασία διαθεσμική για το θέμα αυτό, μια ομοφωνία θα έλεγα, με τους σκιώδεις εισηγητές. Προετοιμάζουμε ένα κοινό ψήφισμα από όλες τις πολιτικές ομάδες, ελπίζω τουλάχιστον, έτσι ώστε να υιοθετηθεί μια κοινή στρατηγική η οποία θα βασίζεται στις αρχές που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί σαν βασικές προϋποθέσεις, όρους, έτσι ώστε στο τέλος της διαδικασίας να στηρίξουμε το κείμενο αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό ε, είναι να ακουστεί βεβαίως και η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτό το πακέτο PNR, αλλά και να ακούσουμε και τα διάφορα συνταγματικά δικαστήρια που πρέπει να σας πω ότι περιμένουν και ελέγχουν πάρα πολύ προσεκτικά όλα τα νομοθετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συντομότερο δυνατόν λοιπόν θα πρέπει ε, ενδεχομένως στην Ολομέλεια του Απριλίου να στηρίξουμε και να υιοθετήσουμε αυτό το κοινό ψήφισμα και πραγματικά κάνω μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να επισπεύσει τις εργασίες της και κατά κάποιο τρόπο να επισπεύσει και όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία. Θα προσπαθήσω να είναι έτοιμο το κείμενο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα ήθελα επίσης να πω ότι απογοητεύτηκα καθότι δεν μπορέσαμε να έχουμε έτοιμη την έκθεση της Επιτροπής η οποία είναι έτοιμη από το 2004. Υπάρχουν δύο κοινέ, αν θέλετε, αναθεωρήσεις, το 2005, το 2010. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ θετικό αν είχαμε το κείμενο αυτό έτοιμο εδώ και μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Όσον αφορά τις συμφωνίες με τον Καναδά και με την Αυστραλία και την εφαρμογή τους, πιστεύω ότι και στις χώρες αυτές υπάρχει 100% συμμόρφωση και βεβαίως εδώ χρειαζόμαστε λίγο περισσότερες πληροφορίες για τα νέα μέτρα ασφαλείας που έχει προτείνει το Υπουργείο Εσωτερικών στις Ηνωμένε Πολιτείες όσον αφορά τον έλεγχο των επιβατών αλλά και την χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω επιγόντως από το Συμβούλιο να μας δώσει απαντήσεις Όσον αφορά τα ερωτήματα που θέτει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2008, του Νοέμβριου του 2008, υπήρχε τότε μια πρόταση ευρωπαϊκή, αυτή σήμερα δεν υφίσταται πλέον, αλλά στο ψήφισμα εκείνο του 2008 υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα για την χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων. Επίσης τα περίφημα στοιχεία API, Ζητώ λοιπόν από το Συμβούλιο να μας δώσει τις πληροφορίες αυτές που ζητάμε από το 2008, το συντομότερο δυνατόν, ό,τι προτάσεις και να υποβάλει η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη και την προστασία που προβλέπεται από το πλαίσιο για τα δεδομένα στα υπερατλαντικά ταξίδια. Ζητάμε εδώ σαφώς και από την Επιτροπή να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το νομικό καθεστώς της συμφωνίας με τον Καναδά. Από ό,τι μου είπαν, προς το παρόν, μονομερός μόνο υπάρχει ανταλλαγή στοιχείων με τον Καναδά είτε ισχύει είτε δεν ισχύει η συμφωνία, νομίζω ότι αυτή η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ δυσάρεστη, καθότι δεν υπάρχει ε, καμία βεβαιότητα. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ε, ευχαρίστησή μας όσον αφορά τη στήριξη διάφορων ε, φορέων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Έχουμε πληθώρα πληροφοριών που έρχονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά βεβαίως δεν θα πρέπει να μας κατακλείσουν με πληροφορίες, προτάσεις και γνωμοδοτήσεις, καθότι και εμείς χρειαζόμαστε γαλήνη για να μπορέσουμε να εργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Πολλές ερωτήσεις ακούστηκαν και προτάσεις την Προεδρία της Επιτροπής μας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή αλλά και στην Προεδρία. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο από την Επιτροπή, η κυρία Βέρκλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε και το λόγο για λίγα λεπτά. Όπως είπα, και προηγουμένως ε, χαιρετίζουμε την ιδέα που κατέθεσε η συγγήτρια για να αναβάλουμε τις δύο συμφωνίες και να δούμε μια πιο συνολική προσέγγιση. Ε, έχουμε σημειώσει επίσης και την έκκληση για ένα ενιαίο σύνολο αρχών για τα δεδομένα PNR και για την εξωτερική μας πολιτική αλλά και για την εσωτερική μας ε, χρήση. Μας ικανοποιεί λοιπόν πολύ το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να υιοθετήσει ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό τον Απρίλιο, διότι αυτό θα βοηθήσει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορέσει να εξετάσει πιο επισταμένα τα κριτήρια τα οποία θέλει να τηρούνται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατόπιν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κριτήρια όταν θα ε, δημιουργήσουμε τα διάφορα μας μέσα. Είτε θα είναι ένα πακέτο PNR το οποίο θα ε, περιλαμβάνει και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη χρήση δεδομένων ε, επιβατών για εξωτερική χρήση ή και η πρόταση για ένα νέο σύστημα PNR. Όπως είπαμε και προηγουμένως, όσο περισσότερη συνοχή έχουμε, τόσο το καλύτερο. Αλλά καλό θα ήταν να γίνει το, το δυνατόν συντομότερο και να έχουμε και μια σαφή ένδειξη από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μα ικανοποιεί λοιπόν ιδιαίτερα το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δραστηριοποιείται και ετοιμάζει ένα τέτοιο κείμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τη προκειμένου να εργαστεί όσο το δυνατόν συντομότερα και να επιτύχει τη συμφωνία εντό Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα διάφορα μέσα που μόλι σα ανέφερα. Μπορεί βέβαια να καθυστερήσει λίγο ακόμα το θέμα αυτό. Θα πρέπει να δούμε και διευκρινήσεις ε, και τα χρονοδιαγράμματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να επανέλθουμε στο θέμα αυτό αργότερα. Μόλις μου υπενθύμησε η συνάδελφος ότι θα πρέπει να πω και κάποια λόγια για κάποια πράγματα για την έκθεση την οποία ε, ετοιμάσαμε για τη συμφωνία PNR. Είχαμε ενημέρωση και από το γραφείο της Επιτρόπου Μάλστροπ ότι η έκθεση θα αποσταλεί από το γραφείο της στο Κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες, πολύ πριν από την ε, Ολομέλεια του Απριλίου. Επομένως, ε, λογικά θα το λάβετε τις επόμενες μέρες, ε, μπορεί και αύριο ή την Παρασκευή το αργότερο. Το αργότερο στο τέλος της εβδομάδας, λέει ο Μιλήτρια. Ευχαριστώ. Η Προεδρία θέλει το λόγο. Ο κύριος Αγγιλέρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω και την άποψη της Προεδρίας για το θέμα αυτό, για το ζήτημα που συζητάμε αυτό που θα πρέπει να πω εδώ στην Επιτροπή σας ε, είναι ότι προς το παρόν δεν έχει γίνει πολιτική συζήτηση στο Συμβούλιο, διότι είμαστε εν αναμονή των περισσότερων λεπτομεριών από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, παρακολουθούμε στενά το θέμα, έχουν υπάρξει επαφές ε, για να είμαστε ενημερωμένοι και να προετοιμάσουμε και το έδαφος αυτή τη στιγμή λάβουμε τη θέση σας ε, για να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να προωθήσουμε τη συζήτηση η οποία λογικά θα μας επιτρέψει να υιοθετήσουμε και μια πολιτική θέση επί του θέματος. Έχουν γίνει βέβαια ανταλλαγές απόψεων με τα κρατημέλη στα πλαίσια των ομάδων εργασιών και οι προκαταρκτικές αντιδράσεις που είχαμε για την τοποθέτηση της Επιτροπής σας είναι θετικές. Θετικές ε, καταρχάς για τη ρεαλιστική τοποθέτηση που ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην έχουμε ένα νομικό κενό το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και πολύ σημαντικές ε, συνέπειες για τους Ευρωπαίους αερομετοφερείς και όπως σας είπα ως πρώτη προκαταρκτική αντίδραση θεωρείται ότι είναι θετικό το γεγονός ότι διατηρείται το status quo στις ε, υφιστάμενες συμφωνίες και προσπαθούμε να προχωρήσουμε λίγο σε αυτή τη ε, διαθεσμική συνένεση τόσο για τις εξωτερικές συμφωνίες αλλά και για την υιοθέτηση ενός εσωτερικού PNR Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπάρχουν κάποιες ιδέες οι οποίες παρουσιάστηκαν στην ε, Προεδρία ε, όπως σας λέω σε επίπεδο προκαταρκτικό δεν είναι οριστικό τελειωτικό το επίπεδο, το πολιτικό επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται αποφάσεις αλλά είναι κάποια ένδειξη. Οι υφιστάμενες ε, συμφωνίες για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να υπάρχουν ε, συγκεκριμένε θέσεις ε, είναι διαφορετικές χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο λαμβάνει θέση μόνο για μία ή για άλλη. Το πιο σημαντικό θα ήταν να έχουμε μία κοινή θέση, αλλά αυτή τη στιγμή καθοριστούν αυτές οι συγκεκριμένες αρχές, τα κριτήρια, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διάφορες καταστάσεις και τα διάφορα πλαίσια στα οποία έχουν επιτευχθεί οι συμφωνίες. Ένα σημαντικό μήνυμα είναι ότι πολλά κράτη-μέλη εμένει στην ανάγκη υιοθέτηση ενό συστήματο PNR στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω γνωρίζετε πολύ καλά εσεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει συζητηθεί και συζητάται εδώ και δύο χρόνια μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία απόφαση πλαίσιο η οποία ε, δεν ισχύει πλέον με την έναρξη ισχύω της συνθήκης της Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια πρόταση επιτάπητος, αλλά όπως ε, είπαμε υπάρχει ε, η συνειδητοποίηση από πλευράς όλων ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να υιοθετηθεί αυτό το σύστημα μέσω μιας νομοθετικής πρότασης που θα πρέπει να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όπως γνωρίζετε αυτό έχει συμπεριληφθεί μεταξύ των προτεραιοτήτων του προγράμματος της Οχόλμης που υιοθετήθηκε στο τέλη του έτους. Αυτά μπορώ να σας πω προς το παρόν. Όσον αφορά στην εξέταση των συμφωνιών αυτών, το Συμβούλιο είναι εν αναμονή και πάλι της ε, κοινή αναθεώρησης της συμφωνίας PNR με τις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον προηγούμενο μήνα και ελπίζουμε να δημοσιευθεί ή να διαβιβαστεί σύντομα. Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι είμαστε θετικά διακείμενοι σε αυτή την πρόταση να έχουμε μια κάποια συνοχή Ελπίζουμε να υιοθετηθεί αυτό το ψήφισμα, στο οποίο το Κοινοβούλιο θα καθορίσει κάποιε βασικέ αρχέ και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι αυτό θα αποτελέσει το εφαλτήριο για αυτή την κοινή ε, τοποθέτηση για τι προτάσει που θα πρέπει να παρουσιάσει στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίε θα επιτρέψουν ε, και στο Συμβούλιο να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση ε, και τη συζήτηση ή να υλοποιήσει αυτέ τι προτάσει να υπενθυμίσω ότι το PNR το ευρωπαϊκό ε, θα προκύψει από συναπόφαση ε, βάσει και τις, τα όσα, των όσων ισχύουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την Προεδρία και τώρα... Υπάρχει σαφή πρόταση τη κυρία Σίνεντφιλτ να αναβληθεί η ψηφοφορία στο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο περαιτέρω την ε, θέση του Κοινοβουλίου, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη των μελών της Επιτροπής μας. Ο κύριος Βος. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια καταρχάς για τη συνεργασία, έξοχη συνεργασία και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Στην ουσία τώρα, συμφωνώ απολύτως με την πρόταση αναβολής για διάφορους λόγους. Αφενός, Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που ίσως θα ήταν βεβαιασμένες. Ε, αυτό σημαίνει ότι αποφεύγουμε τις συνέπειε. και το θέμα είναι να μην υπάρξουν κενά όσον αφορά την ασφάλεια. Αλλιώς η προστασία των δεδομένων θα πρέπει να μας αφήσει εδώ στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να υποβάλουμε τη δική μας, αν θέλετε, θέση, δηλαδή κατά την μεταβίβαση στοιχείων σε τρίτες χώρες, να υπάρχει μία θεσμοθετημένη και ξεκάθαρη διαδικασία, να δώσουμε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε τη δυνατότητα Εάν υπάρξουν ε, κάποια αιτήματα συγκεκριμένα όπως αυτά που έχουμε εδώ ή κάποια άλλα που θα προκύψουν στο μέλλον, να έχουμε, αν θέλετε, ένα πρότυπο, ένα μοντέλο για αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε αυτό να ισχύει για όλες τις μελλοντικές περιπτώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν. Ίσως, λοιπόν, τον Απρίλιο, όταν ε, είμαστε σε θέση να πάρουμε αυτή την απόφαση. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα βασικά προβλήματα, όπως παραδείγματο χάρη οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να μας πούνε τι ανάγκες υπάρχουν, ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες που πρέπει να μεταβιβάζονται και τι ακριβώς είναι, αν θέλετε, αυτά τα δεδομένα αυτά τα στοιχεία PNR επιπλέον όλων αυτών που μεταβιβάζονται. Ε, και εμείς και το Συμβούλιο και η Επιτροπή ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε τη δυνατότητα να αναβληθεί το θέμα αυτό, να μην πάρουμε δηλαδή την απόφαση τόσο σύντομα, γιατί πραγματικά αυτή η προστασία των δεδομένων είναι ένα πιο γενικό θέμα και εμείς σαν Κοινοβούλιο έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για μένα η πρώτη μου αντίδραση όσον αφορά την αναβολή δεν είναι πάρα πολύ θετική. Κοιτάω όμως εδώ αυτό το θέμα το συγκεκριμένο των στοιχείων PNR και πιστεύω ότι όντως υπάρχουν κάποιοι λόγοι να μην βιαστούμε να πάρουμε την απόφαση. Άρα υπάρχουν κάποιοι λόγοι για αναβολή. Χρειάζεται ενδεχομένως μία νέα εντολή και η απόφαση αυτή βεβαίως δεν μπορεί να αναβάλλεται επάπειρον. Ποια είναι τα στοιχεία, για ποια δεδομένα μιλάμε Αυτά τα ξέρουμε. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί, αλλά η εισηγήτρια νομίζω προτείνει τον Απρίλιο. Μέχρι τον Απρίλιο, την Ολομέλεια του Απριλίου, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε. Γνωρίζουμε το θέμα αυτό της συμφωνίας για τα δεδομένα PNR. Και ναι, εντάξει, αν υπάρχουν επιπλέον λόγοι να αναβληθεί αυτή τη στιγμή η ψηφοφορία θα το δεχτούμε, αλλά είναι επίγον το θέμα, η προστασία των δεδομένων, για ποιο λόγο, για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία η αρχική, αν θέλετε, δικαιολογία ήταν η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σήμερα ξέρουμε ότι δεν είναι αυτό το επίκεντρο, αν θέλετε, του θέματος αυτού. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ξεκάθαρα για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία και με ποιο τρόπο το θέμα δεν είναι καινούριο, η συζήτηση δεν είναι καινούρια και πιστεύω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα πρέπει να προχωρήσουμε και να πάρουμε μια απόφαση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα πολύ συγκεκριμένα να πω ότι το θέμα αυτό των προσωπικών δεδομένων των επιβατών λειτουργεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν οι αεροπορικές εταιρείες οι οποίες έχουν τα στοιχεία αυτά και από εκεί και πέρα η πρόσβαση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη για όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Και κανείς ε, δεν μπορεί εδώ να πει συγκεκριμένα ποιο πρακτορείο, ποια αεροπορική εταιρεία, ποια εθνική αρχή, ποιος οργανισμός έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Ακριβώς γι' αυτό το σύστημα αυτό συλλογή στοιχείων ε, για τους επιβάτες δεν ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή στα δεδομένα και στις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι δεν είναι ξεκάθαρο ποια δεδομένα επεξεργάζεται το σύστημα και για ποιο σκοπό. Αυτό είναι πολύ, ε, αν θέλετε, συγκεκριμένο που σας λέω και ενδεχομένως και ε, οργανωμένοι εγκληματίες και τρομοκράτες θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, είτε να τα τροποποιήσουν είτε να τα επεξεργαστούν. Έχω την εντύπωση ότι η αξιολόγηση αυτών των στοιχείων δεν νομίζω ότι είναι περιορισμένη και πραγματικά όταν μιλάμε για καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν νομίζω ότι προστατευόμαστε μέσω αυτού του συστήματος. Η Επιτροπή μας υποσχέθηκε μια νέα πρόταση και πιστεύω ότι η πρόσβαση είναι το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και οι συμφωνίες, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πολύ συγκεκριμένα το άρθρο 8 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Χάρτας, δεν τηρούνται εδώ. Δεν γίνονται σεβαστά. Και θα ήταν πολύ πιο σωστό αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψει αυτή τη συμφωνία. Δεν θέλουμε όμως να αναλάβουμε αυτήν την ευθύνη, αν θέλετε, να παίξουμε αυτόν τον ρόλο και επειδή θέλουμε να παίξουμε το ρόλο μας στην διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Επουδενή λόγο όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα δεχτούμε μια παράνομη κατάσταση. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια κατάσταση που αντιβαίνει των συμφωνιών. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέα συμφωνία με πολύ υψηλά, αν θέλετε, επίπεδα προστασίας και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εγγύσεις και χρειάζεται αναδιαπραγμάτευση, νέα εντολή και το Κοινοβούλιο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να στηρίξει μια τέτοια συμφωνία, δεν μπορεί να στηρίξει μια τέτοια εντολή από τη στιγμή που βλέπουμε να παραβιάζονται με αυτόν τον τρόπο αυτές οι αρχές. Δεν είναι δυνατό να το δεχτούμε. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι θεμελιώδεις αρχές παραβιάζονται, αγνοούνται επειδή απέναντί μας ο συνομιλητής μας είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη στρατηγική, την οποία προτείνει η συγκεκριμένη Σοφή Ντεφέλτ, δεν χρειάζεται να χάσουμε πολύ χρόνο γιατί όπως έχω ήδη πει σε άλλη ευκαιρία συμφωνώ με τη στατικική της. Νομίζω πως είναι λογική αν θέλουμε να μιλήσουμε βεβαίω σοβαρά με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο θα πρέπει να τους δώσουμε κάποιο χρόνο για να κάνουν αυτό που πρέπει και χωρίς βεβαίω να ε, βλάψουμε ούτε τις αεροπορικές ούτε τους πολίτες. Συμφωνώ λοιπόν με τη στρατηγική και με την πορεία που προτείνει η Σόφι Ιντφέλτ και πιστεύω πως και πάλι σε αυτή τη στρατηγική και πίσω από πολλές παρεμβάσει που ακούσαμε είναι η ιδέα αυτής τη Επιτροπής ότι δηλαδή κάνουμε τα πράγματα όχι ε, βήμα-βήμα αλλά κάνουμε το αντίθετο. Δηλαδή αν έχουμε ένα πρόβλημα με τις τράπεζες και τις, ε, τα εμβάσματα ασχολούμαστε με αυτό. Αν έχουμε πρόβλημα με τις αεροπορικέ εταιρείε και τα στοιχεία των επιβατών συζητούμε με τις, με αεροπορικές εταιρείε και έπειτα με τι ΕΠΑ. Ε, έχουμε μια βάση διμερή, συγκεκριμένη σχέση. Αλλά εφόσον αυτό γίνεται, γιατί όχι εμείς να μην έχουμε τα ίδια προϊόνεκτήματα με τους ε, Αμερικανούς. Και αργότερα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να συζητήσουμε με χώρες που χρησιμοποιούν αυτό το άνοιγμα πρόσβασης στα ευρωπαϊκά στοιχεία ε, ως ε, μοχλό για διμερείς εμπορικές σχέσεις. Πιστεύω λοιπόν και έπειτα αυτό που έχουμε εδώ το είπε η Επίτροπος Ρέντινγκ ότι θα κάνει μια αναθεώρηση όλων αυτών για να αφαιρέσει βασικές γενικές αρχές που δεν προέρχονται από πολιτικές αρχές αλλά από μια θεσμική πρατική και από νομοθεσίες που είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσουμε από, την, από τις αρχές για να φτάσουμε σε πολιτικές θέσεις. Γιατί διαφορετικά μιλάμε για τεράστιες βάσεις δεδομένων. Λειτουργούμε σε ένα πολιτικό κενό, όχι σε νομικό κενό, αλλά σε πολιτικό κενό. Αυτό που είπε πριν από λίγο ο Άλμπερτ είναι σωστό. Ότι χρησιμοποιούν, λέει, αυτά τα στοιχεία για να καταπολεμούν το έγκλημα. Αλλά η κλοπή της ταυτότητας είναι ένα έγκλημα όλο ένα και πιο συχνό και δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για το πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται αυτό ας πούμε με τις τράπεζες, αλλά οι τράπεζες δεν λένε πόσες φορές συμβαίνει να κλαπεί η ταυτότητα των πελατών της, τους, γιατί προφανώς είναι εις βάρος τους. Και άρα μπορεί να φτιάχνουμε εμεί βάσει δεδομένων γιατί δήθεν θα καταπολεμήσουμε το τάδε είδος ε, εγκλήματος, αλλά από την άλλη πλευρά ανοίγουμε την πόρτα για ένα σωρό άλλα, άλλων ε, τύπων εγκλήματα. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη φάση που έχουμε μεγάλες κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές θα πρέπει να δούμε και να καλύψουμε το κενό ε, και την βάση. Δεν έχουμε ε, νομοθετική πρωτοβουλία για να κάνουμε ένα τέτοιο έγγραφο βάσης εμείς, ένα νομικό κείμενο. Μέσα στα κείμενα εδώ της, της προτάσεις της ε, Sophie υπάρχουν αρχές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το κατά πόσο ας πούμε είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο push και όχι pull. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε και για το SWIFT και για το PNR και για άλλου είδους. Τώρα, αν είναι Ε, δυνατότητες για να χρησιμοποιήσουμε το YouTube, το email για τέτοιους σκοπούς ας πούμε, όλα αυτά είναι δυνατά γιατί όλα αυτά βοηθούν στην καταπολέμηση των εγκλημάτων. Θα πρέπει λοιπόν να αναλυφθεί σοβαρά υπόψη μας, υπόψη, η άποψή μας από την Κομισιόν, ώστε να συζητήσουμε τις βασικές αρχές και κατά προτίμηση να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και με το Σύνταγμα για να προωθηθούν τα βασικά δικαιώματα προστασίας δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Και εδώ θα μπορέσουμε έτσι να διαπραγματευτούμε με την ίδια σαφήνεια προθέσεων και νομικής ε, βάσης και έτσι θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε επί ίσης με την Αμερική, με την Κίνα και με τη Σαουδική Αραβία και όχι να πηγαίνουμε και να διαπραγματευόμαστε με έναν έναν ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόγκς. Σίγουρα είναι πολύ ε, ανόητη η ερώτησή μου, αλλά πριν προχωρήσουμε με την ε, Αυστραλία, πριν μάλλον πάει κανείς στην Αυστραλία, η αεροπορική εταιρεία απαιτεί θεώρηση ή εν πάση περιπτώσει ηλεκτρονική θεώρηση. Άρα έχουν τις πληροφορίες. Γιατί θέλουν δυο φορές τις ίδιες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις. Δεν έχει σηκώσει κανείς άλλος το χέρι του. Ωραία. Ας επανέλθουμε στην εισηγήτρια. Αλλά ίσως πρώτα η Κομισιόν και η Προεδρία θέλουν να αντιδράσουν στα σχόλια που έγιναν πριν να στραφούμε στην ε, εισηγήτρια. Όχι. Ωραία. Η εισηγήτρια, κυρία Ιντφελτ. Αυτή ήταν ε, η πιο κεντρική και κέρια ερώτηση. Καθόλου ανόητη δεν ήταν και θα ξεκινήσω με αυτήν είναι ένα από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από το Συμβούλιο. Τα ερωτήματα που ανέκυψαν στο ε, περίφημο ψήφισμα του Νοεμβρίου του 2008. Και να πούμε για άλλη μια φορά, στο Συμβούλιο ιδιαίτερα, αυτό που χρειαζόμαστε εδώ χρειάζεται να αποδείξετε την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα όχι απλά την χρησιμότητα των στοιχείων PNR, μα την αναγκαιότητα μαζικής συλλογής και αποθήκευσης των στοιχείων. Δεν μιλάμε για χρήση στοιχείων PNR επί τη βάση ενός εντάλματος σε συγκεκριμένες υποθέσεις, αλλά μιλάμε για την μαζική συλλογή και αποθήκευση στοιχείων χωρίς ένταλμα. Περί αυτού μιλάμε. Και πρέπει να αποδείξουμε την ανάγκη της χρήσης στοιχείων PNR πριν από τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη για τον εντοπισμό των ανθρώπων, την ταυτοποίηση των ανθρώπων. Τα στοιχεία PNI είναι στοιχεία συμπεριφοράς, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν Ε, για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση ανθρώπων είναι στοιχεία συμπεριφορά. Ε, αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκεί είναι τα στοιχεία APA, Advanced Passengers, ε, Passenger Information. Αυτά είναι μόνο στοιχεία που δίνουμε στο σύστημα κρατήσεων όταν κλείνουμε ένα εισιτήριο. Και άμα θέλω να βγάλω εγώ εισιτήριο στο όνομα του Mickey Mouse, μπορώ. Αν δείτε, πώς, δείτε και πώς γράφεται το όνομά μου και στην ατζέντα σήμερα για τη σημερινή συνεδρίαση, λάθος το έχουν γράψει και πάντα το γράφουν λάθος. Σας το εγγυώμαι ότι ακόμα και η οικογένειά μου ανάμεσά μας τσακωνόμαστε πώς γράφεται σωστά το όνομά μου. Άρα λοιπόν τα στοιχεία PNR δεν χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. Χρειάζεται δηλαδή να αποδειχτεί η αναγκαιότητα και όχι μόνο σε εμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να σας το θυμίσω αυτό. Θα πρέπει να το αποδείξουμε, να αποδειχτεί μάλλον και στα διάφορα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια. Να, να πείσουμε δηλαδή το συνταγματικό δικαστήριο δικαστρούης ότι αυτό είναι αναλογικό. Και άμα νομίζετε ότι εγώ είμαι σκληρή, αυτή είναι χειρότερη. <coughs> Για την πρόταση αναβολής. Όπως ε, και η κυρία Ήπολ ε, και ο Άλμπρεχτ, ε, δουλεύω για αυτό το θέμα από το 2004, προκάτοχός μου από το 2003. Αν με ρωτούσατε αν θέλετε να ψηφίσουμε σήμερα και να το απορρίψουμε τελείως, ε, ναι, πολύ θα το ήθελα. Βλέπω, με κοιτάζει με ορθάνυχτα μάτια ο κύριος Μπουσουτήλ, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν ανεύθυνο κάτι τέτοιο ότι θα ήταν πολύ πιο επικοδομητικό να προσπαθήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε την κατάσταση για να φτάσουμε σε μια πολύ καλύτερη λύση. Ε, να θυμίσω στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν που είναι νέοι σύμμαχοι σε αυτή την υπόθεση ότι το θέμα δεν έχει φύγει. Γι' αυτό και συμφωνώ με την κυρία Ζήπελ ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα η πρόταση. Ολοκληρωμένη, η πρόταση υψηλής ποιότητας, αλλά και ταχύτατα και μια τελεκυφταία πρακτική παρατήρηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει κυκλοφορήσει ευρέως το ψήφισμα γιατί θεωρώ πως είναι θέμα ευγένεια στους και ηγητές να συμφωνήσουμε για ένα κείμενο πριν κυκλοφορήσει. Ξέρω ότι ορισμένοι άλλοι ε, διαφωνούν, αλλά δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει σίγουρα πριν να έχουμε συμφωνήσει για ένα κείμενο. Μόλις θα έχουμε συμφωνήσει, σας διαβεβαιώ πώς θα το λάβετε, γιατί πιστεύω πως θα μας βοηθήσει κάτι τέτοιο ώστε να φτάσουμε σε θετική ψήφο τον Απρίλιο. Ευχαριστώ κυρία Άινελβελτ. Ποτέ δεν είμαι βέβαιος αν προφέρω το όνομά σας σωστά. Mm. Πώς προφέρετε, είναι Τέλος πάντων λίγο πολύ το βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι υπάρχει συνένεση για την πρότασή σας. Να αναβάλουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Όλα τα μέλη και όλες τις πολιτικές ομάδες που εξέφρασαν την άποψή τους συμφωνούν και νομίζω ότι Ολοκληρώσαμε για σήμερα γιατί έχουμε καλύψει τα σημεία που είχαμε για την απογευματινή συνεδρία της Επιτροπής μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αύριο το πρωί στις 10. Αύριο στις 10. Για τη συνεδρίαση αύριο ψηφίζουμε. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν να φέρετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Ευχαριστώ πολύ.